2 Απριλίου 2014 θα ανήκει στους μη εγγεγραμμένους. Από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχω κάποια αιτήματα για διορισμού σε αντιπροσωπείες και διακοινοβουλευτικές ε, επιτροπές. Θα δημοσιευθεί στα πρακτικά. μέχρι την δημοσίευση αυτή ε, δεν θα υπάρχουν στάσεις, θεωρείται ότι κυρώνεται αυτός, κυρώνται αυτοί οι διορισμοί. <clears throat> και σύμφωνα με το αρμόδιο άρθρο έχουμε 34, 34 νομικές πράξεις που έχουμε υπογράψει με τον πρόεδρο